Καθίστε παρακαλώ γιατί θα ξεκινήσουμε με το σημείο υπαριθμών 14 ανταλλαγή απόψεων με τον ε, κύριο Γκαρίγα Πογέδο για την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ που είναι η Επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με τις ε, δαπάνες και τις ε, πολιτικές πολιτή χρηματοδότηση μετά το 2013. Ο κύριος Πογέδο είναι ο εισηγητή για την Επιτροπή Σούρα και ανήκει στην Επιτροπή Προπολογισμών και θεώρησα ότι είναι καλό να έρθει να μα ε, ε, μιλήσει γιατί άλλωστε η πρόεδρο τη προσωρινής επιτροπής ζήτησε συνεργασία με όλε τι ε, ε, επιτροπές. Να σας πω επίσης ότι ο υπουργό των Εξωτερικών του Νησιών Φερόε θα έρθει όπου να είναι και μόλις έρθει θα σταματήσουμε την ενημέρωση από τον κύριο Γκαρίγα Πογέδο και θα ακούσουμε τον Υπουργό και θα συνεχίσουμε αργότερα. Ε, να δώσω όμως το λόγο στον κύριο Γκαρίγα μέχρι να έρθει ο υπουργό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Αλληλείας, όπως επίσης και η γνωμοδότηση των άλλων επιτροπών, θα είναι ιδιαίτερο χρήσιμη όταν θα ξεκινήσουμε την τομεακή ανάλυση για τις επόμενες δημοσιονομικές προπτικές. Και στη συνέχεια θα σας εξηγήσω και λίγο το χρονοδιάγραμμα. Θα ξεκινήσουμε από το Φεβρουάριο. Η Επιτροπή αυτή, η οποία είναι μια προσωρινή Επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τις δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013, έχει την εξή εντολή να καθορίσει τις πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το επόμενο διάστημα των δημοσιονομικών προοπτικών, να υπολογίσει τους δημοσιονομικούς πόρους που απαιτούνται και να καθορίσει και τη διάρκεια του πολιετούς πλαισίου θα υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες, μια συγκεκριμένη δομή, κάποιες κατευθυντήριες ευδικτικέ γραμμές για την ανάθεση των πόρων, και την κατανομή των πόρων και ε, μια ιδέα για τις ε, δαπάνες καθώς επίσης και το θέμα της μεταρρύθμισης του συστήματος χρηματοδότησης του προπολογισμού, διότι συμφωνούμε όλοι ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσουμε την ε, τον προπολογισμό που είχαν συνεισφέρει μέχρι τούδε τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, η συζήτηση θα εστιάσει κυρίως ε, στους απαραίτητου πόρους και τις απαραίτητε δαπάνες. Και φυσικά, ε, σε αυτή τη συζήτηση θα θέλαμε να συμπεριλάβουμε και άλλου δημοσιονομικούς πόρους που θα επιτρέψουν τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει ένα επίπεδο δαπανών το οποίο θα είναι συγκρίσιμο με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, Και ναι, μεν θα είναι χαμηλότερο από τι προηγούμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ, αλλά ε, γενικότερα παρατηρούμε ότι η τάση σε αυτά τα χρόνια τη κρίση για τα κράτη-μέλη θα διατηρηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα. Θα θέλαμε λοιπόν να κάνουμε μία αναθεώρηση των απαραίτητων πόρων. Οι εργασίε μα θα πρέπει να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2011 θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου μία έκθεση με την οποία έκθεση θα προσπαθήσουμε να τηρήσουμε την εντολή που μας έχει δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχουμε το εξή σύστημα εργασίας. Θα καλύψουμε καταρχάς τις βασικές αρχές. Οι βασικές αρχές ε, είναι καταρχάς η σημασία και η προστιθέμενη αξία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν θέλουμε να καθορίσουμε τους ε, δημοσιονομικέ δαπάνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και επίση, αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία τη συζήτηση για τη στρατηγική για το 2020 το πώ θα επηρεάσει αυτό τι δαπάνε και ε, το μέλλον για τις ε, δημοσιονομικέ προοπτικές. Υπάρχει μια άμεση σχέση μεταξύ τη Δομή του 2020 και των επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών αλλά η στρατηγική για το 2020 δεν θα καλύπτει όλα όσα καλύπτουν οι παρούσες δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, βέβαια όσα αφορούν τη δική σας επιτροπή λογικά θα καλύπτονται από εκεί διότι θέλουμε η προηγούμενη κατηγορία 2 να ενσωματωθεί στην ε, στρατηγική για το 2020 και για την άμεση χρηματοδότηση αλλά και για τις διάφορες τομεακές πολιτικές. Και επομένως η αλληλεία θα συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική του 2020. Ε, είτε στον ε, άξονα της ανάπτυξης είτε σε οποιοδήποτε άλλον από τους δύο άξονες. αλλά θέλουμε να έχουμε επαρκή χρηματοδότηση της πολιτικής αλληλείας για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή τώρα θα έχουμε αναλύσει τα διάφορα στοιχεία, παραδείγματος χάρη την προστίθωμενη αξία, την εκτέλεση του προπολογισμού, ε, τι, ακριβώς θέλουμε να έχουμε σε επόμενες ε, δημοσιονομικές προοπτικές θα συμπεριλάβουμε και μία ανάλυση για το τι είναι απαραίτητο για το μέλλον, μία ανάλυση για τους νέους ίδιους πόρους, ε, τα νέα ε, βασικά στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και από το Φεβρουάριο-Μάρτιο θα ξεκινήσει μια διαδικασία ανάλυσης των τομεακών πολιτικών και εκεί η πρόεδρος της Επιτροπής μας, η Γιούτα Χάουγκ, έχει ήδη ε, υποβάλει σχετικό αίτημα στις αρμόδιες επιτροπές για να συμμετέχουν και αυτές στη διαδικασία συζήτησης με την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής αλληλείας και πού θα πρέπει να τοποθετηθεί σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής του 2020 πολιτική αλληλεία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλείας. Θα πρέπει λοιπόν η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή να συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις. Σε αυτή την πρώτη φάση λοιπόν ε, θεωρώ ότι θα εργαστούμε στα πλαίσια της Επιτροπής ε, ΣΟΥΡΕ, θα καθορίσουμε τις βασικές κατευθυντηρίες γραμμές και όταν θα φτάσουμε στις τομεακές πολιτικές θα φτάσει και η στιγμή για την πιο στενή συνεργασία μεταξύ ε, της προσωρινής Επιτροπής και της Επιτροπής Αλίας. Είναι προ το συμφέρον εννοείται των μελών της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ όλες οι αρμόδιες επιτροπές, κυρίως οι επιτροπές που κάνουν έλεγχο ή κατευθύνουν ή δίνουν προσανατολισμούς για τις ε, κοινοτικές δαπάνες να συμμετέχουν στις εργασίες και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ε, ΣΟΥΡΕ. Ε, δεν έχει ακόμα καθοριστεί πώς ακριβώς θα γίνει τη συνεργασία. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εκπονήσει έκθεση η Επιτροπή Αλίας και να την υποβάλει στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ. Το πιο απλό θα ήταν ο εισηγητής της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, δηλαδή εγώ, να συμμετέχω σε κάποιες ε, συγκεκριμένες συνεδριάσεις της Επιτροπής Αλίας. Αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο θα αναλύσουμε κυρία Πρόεδρε στην ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών φαντάζομαι. Αυτά λοιπόν ως γενική εικόνα της κατάστασης αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ και το αίτημά μας για μελλοντική συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Γκαρίγα. Εγώ είχα προβλέψει να έρθετε διότι έχετε διπλή αρμοδιότητα. Είσαστε εισηγητής, όπως ε, μας είπατε, ε, για την έκθεση που θα πρέπει να ετοιμάσει η Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, αλλά επίσης είστε και μέλος ε, της Επιτροπής Αλίας. Επομένω, ελπίζουμε ότι εσείς θα αποτελέσετε το διάβλο για μεγαλύτερη επικοινωνία, διότι θα είστε και λίγο πιο... έχετε μεγαλύτερες ευαισθησίες και θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε στο μέλλον. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού πλαισίου θα συζητηθεί τώρα, αλλά προβλέπετε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα ξεκινά από το 2013 ή θα καθυστερήσει η ισχύ ε, αυτού του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, διότι έχω ακούσει διάφορες ε, απόψεις, δεν ξέρω ποια είναι η θέση της προσωρινής επιτροπής και δεύτερον θα ήθελα να επισημάνω το εξής. συζητάμε μια μεταρρύθμιση. Ε, βέβαια θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει ότι θα γίνει και μεταρρύθμιση της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν σχέση οι δύο μεταρρυθμίσεις μεταξύ των. Δεν θα ανακατευτώ εγώ με τα θέματα της γεωργίας γιατί δεν είναι δική μου δουλειά, αλλά νομίζω ότι η Αλία και η Γεωργία μας εντάσσουν στην ίδια κατηγορία, στην κατηγορία 2 και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να επισημάνω το σημείο αυτό. Η μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής ε, και η χρηματοδότηση που λαμβάνουμε εμείς δεν είναι ούτε καν ε, ένα δις ευρώ. Αν καταλα... το βλέπετε κι εσείς, είμαστε ο τελευταίο τροχός αμάξης. Δεν έχουμε καμία σχέση με την κοινή γεωργική πολιτική, γιατί αυτοί παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμά. Το κόστος λοιπόν της μεταρρύθμισης θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα διακόψουμε τώρα, γιατί μόλις έφτασε ο Υπουργός και μετά θα συνεχίσουμε μαζί σας κύριε Γκαρίγα. Κύριε Γκαρίγα, θα δείχνετε κατανόηση. Επιτρέψτε μου να ακούσουμε λοιπόν τον Υπουργό και να ξεκινήσει το σημείο αυτό και θα συνεχίσουμε μετά. Κύριε Υπουργέ, καλωσορίσατε στην Επιτροπή Αλίας. Όπως ε, γνωρίζετε, η Επιτροπή μας ανησυχεί ιδιαίτερα για τις διαπραγματεύσεις και για την ε, αλία Έχετε πολλά πράγματα να μας πείτε για το Ιναλία στην περιοχή σας. Ε, ε πέραν από την πρόσκληση σε εσά. Έχουμε απευθύνει πρόσκληση και στην Υπουργό τη Ισλανδία και ε, δυστυχώ βέβαια λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να έρθει. Ξέρετε ότι υπάρχει αρμόδιος εισηγητής ε, ο οποίος ενδιαφέρεται όχι μόνο γιατί είναι Σκοτσέζος αλλά γιατί ε, τον ενδιαφέρει και το θέμα και είναι και δήμον επί του θέματος ε, και έχει έρθει σε επαφή μαζί σας. Στη συνέχεια λοιπόν της συνεδρίασής μας θα μπορέσετε να μας πείτε κάποια πράγματα για το Σαφρίδι διότι γνωρίζετε και εσείς κάποια πράγματα και για το πόσο μας ενδιαφέρει και ε, νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να ακούσουμε και το μέλη της Επιτροπής που θα μπορέσουν να σας θέσουν ερωτήσεις. Καλώς ορίσατε. Ε, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ και σας δίνω το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα ευχαριστώ να, καταρχήν να ευχαριστήσω την πρόεδρο της Επιτροπής την κυρία Κάρμεν Φράγα Εστέβες για την πρόσκληση που μου απέστειλε για να μιλήσω σήμερα στην Επιτροπή σας. Είναι μια ευκαιρία για μένα για να παρουσιάσω τις απόψεις μας ενώπιόν σας για τη διαχείριση του σαφριδιού στο βορειοανατολικό Ατλαντικό. Χαίρομαι, χάρηκα επίσης για τη χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων που είχα τον περασμένο μήνα στα νησιά Φαρόε με την με τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Στρούαν Στίβενσον και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω που ε, ανέλαβε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί αυτή η συζήτηση. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα νησιά Φαρόε, σε ένα ανοιχτό διάλογο και σε μια ανταλλαγή πληροφοριών. Πιστεύουμε ότι είναι ο ακρογωνιαίος λήθος της συνεργασίας μας στον τομέα της Αλίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους εταίρους στο Βόρειο Ατλαντικό. Ο συνάδελφός μου, ο Γιάκομπ Φέστεργαρντ, ο Υπουργό Αλίας των νήσων Φάροε, είναι υπεύθυνο για τη συμμετοχή των νησιών στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των παρακτήων κρατών και της... Και υπεύθυνο επίσης για τη διαχείριση της αλίας στα νησιά Φαρόε εν γέννη. Θα ήθελα επίση εκ μέρου να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή και μου ζήτησε να τον εκπροσωπήσω επίσης σε αυτή τη συνάντηση. Τώρα, για το θέμα που μας απασχολεί σήμερα, δηλαδή η κοινή διαχείριση του σαφριδιού. Θα ήθελα να πω ότι αισθανθήκαμε περίεργα και αισθανθήκαμε έκπληξη από τον επιθετικό τρόπο με τον οποίο το θέμα περιγράφτηκε τις πρόσφατες εβδομάδες, όχι μόνο στα ΜΜΕ, αλλά και εδώ, στο επίσημο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατήρησα ότι αυτή η επιτροπή, η σας αναφέρεται στο θέμα αυτό ως μία διαμάχη με τα νησιά Φαρόε και με την Ισλανδία και αναφέρεται στα μέτρα διαχείρισής μας του 2010 ως απαράδεκτα μέτρα και απαράδεκτη συμπεριφορά. Είναι σαφές, κατά την άποψή μου, ότι πρέπει να πάμε λίγο πίσω για να δούμε που, πώς στάσανε οι συζητήσεις εδώ και να δούμε, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα πιο ισορροπημένα και με μια προοπτική. Γι' αυτό λοιπόν ε, χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία για να σας δώσω κάποια στοιχεία και να σας πω ποια είναι η προοπτική ε, που έχουμε εμείς στα νησιά μας. Τη στιγμή που συναντιόμαστε εδώ, ένας δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων και από τα τέσσερα παράκτια κράτη βρίσκεται να εξελίξει στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος γύρος των συζητήσεων πριν από δύο εβδομάδες ήταν ε, χρήσιμος και προέκυψε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, καθώς και είδαμε ότι υπάρχει επιθυμία από όλα τα μέρη να βρεθεί μια διαρκής λύση. Τουλάχιστον εμείς αυτό προσπαθούμε εργοδός. Ίσως είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο τομέα αλίας. Βλέπετε τα νησιά στο κέντρο του χάρτη. Είμαστε μικρή χώρα, αλλά έχουμε μια κεντρική θέση και ένα κεντρικό ρόλο στην ε, συνεργασία στον τομέα της Αλίας στο βορειοανατολικό Ατλαντικό. Είμαστε ένα έθνος το οποίο εξαρτάται πάρα πολύ από την Αλία και αναλογιζόμαστε την ευθύνη αυτή. Επομένως θεωρούμε ότι είναι υποχρέωσή μας να συνεργαστούμε με όλα τα έθνη για τη διαχείριση των κοινών μας πόρων. Και Έχουμε μια μακρά παράδοση θαυμάσιας διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της αλίας στο βόρειο Ανατολικό Ατλαντικό και σε διμερή βάση, αλλά και μέσω των ε, ρυθμίσεων που βρίσκουμε τα παράκτια ε, κράτη, καθώς και με τη συμμετοχή σε περιφερειακούς ε, οργανισμούς όπως η ΝΙΑΦ και η ΝΑΦΕ. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει στενή και επικοδομητική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό συμπεριλαμβάνει τη συνεργασία και για την επιστημονική έρευνα και για τα θέματα του ελέγχου. Ο ωκεανός μας δίνει πράγματα, αλλά μας παίρνει κιόλα. Όπως ανέφερα, η οικονομία των Φαρόε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλία και την υδατοκαλλιέργεια. Αυτό, αυτή η κλάδη στα νησιά στα νησιά μας δίνουν το 95% των εξαγωγών μας και 60 με 70% του συνολικού εισοδήματος από τις εξαγωγές. Επίσης, η αλία είναι πάρα πολύ σημαντική για... και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια δίκαιη κατανομή των, αποθε... των αποθεμάτων, δηλαδή του σαφριδιού, της Ρέγκας και του προσφυγακίου. Αν κοιτάξετε το χάρτη που έχουμε εδώ, να σας κάνω ένα μικρό έτσι τεστ. Έχουμε το προσφυγάκι με μπλε χρώμα, την ρέγγα κόκκινη και κίτρινη, το κίτρινο χρώμα αφορά το σαφρίδι. Πρέπει να δούμε πώς θα ανακατέψουμε αυτά τα χρώματα στην παλέτα. Γιατί το μπλε είναι γύρω-γύρω, το βλέπετε, στα νότια και στα βόρεια μέχρι ψηλά. Η ρέγκα είναι περίπου στην ίδια περιοχή με το κόκκινο και το σαφρίδι ανακατεύεται με τα άλλα χρώματα και μας δίνει ένα πράσινο ή ένα πορτοκαλί ανάλογα. Επομένως, τα περισσότερα από τα πελαγικά αποθέματα στα βορειοανατολικά του Ατλαντικού βρίσκονται στα ύδατά μας, αλλά και γύρω-γύρω. Όλα αυτά τα αποθέματα Ε, υπάρχουν και το καλοκαίρι και επίσης είναι σημαντικό λοιπόν ε, το γεγονός ότι δίνουν τροφή. Τα πελαγικά αποθέματα στα Φαρόε είναι πολύ σημαντικά συνολικά για την αλία μας. Αποτελούν το 40% της αλίας μας σε ό,τι αφορά την οικονομική τους αξία. Τα πελαγικά αποθέματα μιλάω. Αυτό σημαίνει ότι τα νησιά μας ενδιαφέρονται πάρα πολύ να υπάρχει μια κοινή διεθνής διαχείριση των αποθεμάτων. Υπάρχουν δραματικές διακυμάνσεις ε, τα τελευταία χρόνια στη Ρέγα και στο Προσφυγάκι. Βλέπετε και τα νούμερα το δείχνουν αυτό. Ε, Ξαφανίστηκε εδώ και 20 χρόνια περίπου η Ρέγκα αλλά με την διεθνή συνεργασία και τη διεθνή διαχείριση από τα μέσα της δεκαετίας του 90 τώρα είμαστε σε θέση να εποφεληθούμε από ένα υγιές απόθεμα και από μια σχετική σταθερότητα στον τομέα αυτό. Αλλά όμως για το προσφυγάκι δεν έχουμε αντίστοιχες ε, επιτυχίες. Χρειάστηκε πολλής χρόνος για μια τελική συμφωνία και σήμερα υφιστάμεθα τις συνέπειες, γιατί αργήσαμε πραγματικά να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική διαχείριση. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια δίκαιη συμφωνία, συμφωνία για την κατανομή και λαμβάνουμε και προωθούμε κοινέ δράσει ω παράκτια κράτη, ούτω ώστε να μειώσουμε, ε, τουλάχιστον του χρόνου, τα αποθέματα α, δραματικά. Θα ψαρέψουμε πολύ πολύ λιγότερο και πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να, την αποκατάσταση του αποθέματος και τα επόμενα χρόνια η αλληλεία στον τομέα αυτό θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας εμείς στα νησιά μας, γιατί είμαστε αναγκασμένοι και το ξέρουμε. Για πολλά χρόνια το απόθεμα του σαφριδιού ήταν ένα βασικό προϊόν και ένας αξιόπιστος πελαγικός πόρος στην περιοχή μας. Ως τμήμα στην διευθέτηση ατχό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νορβηγία τα 10 χρόνια, τα νησιά Φαρόε ήταν ένας ενεργός συμμετέχων στην κοινή διαχείριση του σαφριδιού. Συνεισφέραμε στην ανάπτυξη του αποθέματος του σαφριδιού ε, και το αποτέλεσμα είναι ότι είναι σήμερα ένα από τα δυνατότερα και πιο πολύτιμα κοινά αποθέματα αλλιευμάτων στον βορειοατλαντικό, στο βορειοανατολικό Ατλαντικό. Τα τελευταία χρόνια είχαμε ένα, ένα ε, εντυπωσιακά μικρό ε, μερίδιο, λιγότερο από 5%. Ένα μερίδιο το οποίο θεωρούμε σήμερα ότι δεν είναι σύμμορφο με μια δίκαιη κατανομή αυτού του πόρου. Με αυτόν τον περιορισμό στη, στα συνολικά αποθέματα του Σαφριδιού στα νησιά Φαρόε δεν μπόρεσαμε να αναπτύξουμε περαιτέρω την αλληλεία. Παρότι υπάρχουν ε, στοιχεία ότι υπάρχει αυθονία Σαφριδιού ε, στην περιοχή μας εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχει βέβαια η κλιματική αλλαγή, αλλά υπάρχει κλιματική αλλαγή και στον ωκεανό. Και όταν υπάρχει κλιματική αλλαγή στον ωκεανό, τα ψάρια μετακινούνται. Και αυτό συνέβη και με το Σαφρίδι. Επομένως θα πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα και θα πρέπει να σκεφτούμε πιο προσεκτικά εν ώψη της κλιματικής αλλαγής. Εμεί θέλουμε να διατηρηθεί η εξαιρετική κατάσταση του αποθέματο του Σαφριδιού και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμείνει το αλίευμα αυτό βιώσιμο στο μέλλον. Αλλά για να το εξασφαλίσουμε αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή για όλους τους συμμετέχοντες και αυτή να είναι η βάση της κοινή μας διαχείρισης. Προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη κατανομή βορειοδυτικά και η αυθονία των χώνων και των ενηλίκων σαφριδιών θα πρέπει να αντανακλάται σε μια νέα συμφωνία κατανομής που να καλύπτει το συνολικό κλάδο της αλίας. Αν κοιτάξετε αυτό το χάρτη θα δείτε πού βρίσκεται το σαφρίδι από το 1980 μέχρι το 2000. Βλέπετε πού κινήθηκε. Τώρα, από το 2000 μέχρι το 2007, βλέπετε ότι το Σαφρίδι μετακινήθηκε βόρεια και δυτικά για τα τελευταία τρία χρόνια, από το 2007 μέχρι σήμερα, πήγε ακόμα πιο βόρεια και ακόμα πιο δυτικά. Και σήμερα τα νησιά Φαρόε είναι το κέντρο της περιοχής όπου ευδοκιμεί το Σαφρίδι. Ενώ πριν 10 ή 20 χρόνια είμαστε πιο περιθωριακοί σε σχέση με το απόθεμα αυτό. Άλλαξαν τα πράγματα στο Βόρειο Ατλαντικό, γι' αυτό χρειαζόμαστε νέα κατανομή. Αυτό σημαίνει μια συμφωνία. Το κοινό οικοσύστημα εποπτεύεται από το Ινστιτούτο που έχουμε στα νησιά Φερόε και το Ινστιτούτο αυτό επιβεβαίωσε ότι η κατανομή και η αυθονία του σαφριδιού είναι πιο βόρεια και πιο δυτικά από ό,τι στο παρελθόν. Βλέπουμε το αποτέλεσμα λοιπόν που είναι το κόκκινο χρώμα. Αυτό σημαίνει περισσότερο σαφρίδι. Ε, λιγότερο σαφρίδι βρίσκεται στο κίτρινο και στο πράσινο χρώμα. Αυτή η μελέτη του Ινστιτούτου δείχνει ότι στα νησιά μας υπάρχουν πάρα πολλά σαφρίδια. Τώρα, για πρώτη φορά τα νησιά συμμετείχαν μέσω του, Ινστιτού, του Θαλάσσου Ινστιτούτου σε μια επιθεώρηση για το Σαφρίδι που γίνεται κάθε τρία χρόνια. Η επιθεώρηση αυτή επιβεβαίωσε ότι επίσης το Σαφρίδι αναπαράγεται στα νησιά μας. Και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα της μελέτης της επισκόπησης του 2007. Με όλα αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας πιστεύουμε ότι τα νησιά Φαρόε έχουν δικαίωμα να αυξήσουν το μερίδιο του στη νέα συμφωνία για το Σαφρίδι. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία της ε, συμφωνίας ad hoc, τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά, τουλάχιστον για μας. Όπως το χάρη η μονομερής κατανομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ε, ενός λεγόμενου νοτίου α, αποθέματος μια νότια συνιστόσα. Ένα είναι το απόθεμα. Επίση, ε, κατά την ρύθμιση αυτή ad hoc, παρατηρήσαμε ότι υπάρχει υποαναφορά των αλλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά είναι μεγαλύτερο από τον νησιών Φερόε. Ορισμένε περιπτώσει περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν επιβληθεί ε, κυρώσει κυρώσεις. Μπράβο σας. Αλλά η ISIS εξακολουθεί να υπολογίζει ότι για το 2010 ε, υπάρχουν ε, υπερεκτιμήσεις ή μάλλον υπάρχουν υπερβολικά μεγάλα αλλιεύματα σαφριδιού. Νομίζω ότι το βάρος είναι κοινό. Όταν στυλιτεύουμε κάποιον, ε, να μην ξεχνάμε ότι μερικές φορές ε, εμείς οι ίδιοι πρέπει να κάτσουμε στο εδόλιο. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μία νέα και πιο διαφανή ε, συμφωνία διαχείρισης του σαφριδιού για όλο το απόθεμα σαφριδιού και που βοηθάει να προωθήσουμε τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο και την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνιών. Δυστυχώς, δεν υπήρχε συμφωνία για το 2010 των παράκτιων κρατών. Το αποτέλεσμα είναι ότι όλα τα παράκτια κράτη, καθώς και η Ρωσική Ομοσπονδία, καθόρισαν ό,τι θεωρούσαν ότι είναι κατάλληλο όριο για, τις δικές τους, για τη δική τους αλία το 2010. Αυτά τα όρια έχουν αναφερθεί στην ΕΑΦΚ με βάση τις συστάσεις για τα διεθνή ύδατα που προσαρμόστηκαν οι συστάσεις αυτές το 2010 τον Ιούνιο συγκεκριμένα. Αλλά η κατάσταση όμως δεν είναι ιδανική. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, καλύτερο αυτό παρά μια αλία εντελώς αρρύθμιστη, εντελώς άναρχη. Τα νησιά Φαρόε αρχίσαμε να ψαρεύουμε σαφρίδι τέλος Ιουλίου. Το Υπουργείο Ελίας στις 23 Ιουλίου ανακοίνωσε την απόφαση να καθορίσει το όριο για το δικό μας απόθεμα σαφριδιού στους 85.000 τόνους. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε και ποσοστώσεις που μεταφέραμε από την Ορβηγία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ρωσία και την Ισλανδία μέσω διμερών συμφωνιών. Αλλά αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνει επίσης και κάποια ποσά που έχουμε θεσπίσει για την επιστημονική έρευνα για την αυθονία του σαφριδιού, καθώς και την κατανομή του στα ύδατά μας. Όλα τα λάβαμε υπόψη μας δηλαδή. Ο λόγος για την καθυστερημένη απόφαση, δεν δηλαδή περιμέναμε μέχρι τις 23 Ιουλίου για να αποφασίσουμε για τα όρια μας, ο λόγος λοιπόν είναι ότι θέλαμε να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Οι διαβουλεύσεις το Μάιο όμως ε, δεν κατέληξαν πουθενά. Εμείς θέλησαμε να προσπαθήσουμε περισσότερο γιατί θέλαμε αυτή τη συμφωνία. Ο Υπουργός λοιπόν Αλίας συναντήθηκε με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και με την Ορβηγία και την Ισλανδία τον Ιούνιο και τον Ιούλιο για να διερευνήσει μήπως υπάρχει ακόμα ευκαιρία για κάποια συμφωνία για το 2010. Αλλά προέκυψε σαφώς ότι δεν υπήρχε υποστήριξη μεταξύ των μερών για να βρεθεί λύση για το 2010. Η αλίευση εντωμεταξύ είχε ξεκινήσει ωραιότατα σε άλλες περιοχές. Το επίπεδο των ορίων για τα νησιά Φαρόε για το Σαφρίδι συνάδει απόλυτα με το επίπεδο του μεριδίου που θεωρούμε ότι είναι δίκαιο για τα νησιά μας με βάση μία μέχρι τώρα στα παράκτια κράτη. Παρά την αργή εκκίνηση έχουμε ψαρέψει όλη την ποσόστοση και η αλία πήγε πάρα πολύ καλά στο, για το σαφρίδι. Μόνο μέσα σε 60 μέρες εξαντλήσαμε την ποσόστοση ψαρέψαμε αυτά τα ποσά. Όχι απλώς ήταν καλή η αλία, αλλά και πάνω από το μισό τα εκατό που εκφορτώθηκαν στα λιμάνια μας ε, ή μεταποιήθηκαν ήταν για ανθρώπινη χρήση. Μία από τις ε, βασικές τροχοπέδες ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία είχαν εδώ και πολύ καιρό υπογράψει μια διμερή συμφωνία μεταξύ του για το Σαφρίδι το 2010 και αυτό φυσικά περιέπλεξε τις διαπραγματεύσεις. Ο συνδυασμένο ε, βαθμός των ποσοστώσεων που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία το 2010 είχαν ξεπεράσει το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα που είχε συστήσει ο ISIS. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η Νορβηγία μετέφερε περίπου 70.000 τόνους Τη μη χρησιμοποιηθή σα που είχε το 2009, τη μετέφερε λοιπόν στο 2010. Αυτές οι μεταφορές δεν ήταν ποτέ τμήμα τη προηγουμενη ad hoc ρύθμιση στην οποία συμμετείχαν και τα νησιά Φαρόε. Αλλά αυτό το ευλόγησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2010, από ό,τι φαίνεται. Ο συνδυασμένο βαθμό ποσοστώσεων Ευρωπαϊκή Ένωση και Νορβηγία δεν άφησαν κανένα περιθώριο ελιγμών για τα υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη για το 2010. Το γεγονός ότι χωριστές μονομερεί ποσοστώσεις καθιερώ, ε, θεσπίστηκαν από όλα τα κράτη ε, που ξεπερνούν το συνολικό επιτρεπόμενο αλήμα δεν είναι κάτι θετικό. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν προκλήθηκε από έναν από εμά. Όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Τα παράκτια κράτη έχουν τώρα μια κοινή ευθύνη για τη διαχείριση του σαφριδιού. Είναι τεσ... Υπάρχουν τέσσερα τα συμβαλόμενα μέρη και η Ισλανδία συμμετέχει πλήρως ως παράκτιο κράτος. Η βασική πρόκληση είναι να ξαναδούμε την προσέγγιση μας και να βρούμε μια νέα ρύθμιση, μια νέα συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων ε, παράκτιων κρατών, ε, φυσικά σε ίση βάση. Όλα τα μέρη έχουν τις δικές τους αξιώσεις και απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους. Εάν τα παράκτια κράτη συνεργαστούν ισότιμα, τότε δεν μπορούμε να εξετάσουμε χωριστά τις απαιτήσεις του ενός και να μην λάβουμε υπόψη μας και τις απαιτήσει των υπολείπων. Όσο και αν είναι δύσκολο, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια νέα κλίδα κατανομής. Μην ξεχνάτε ότι το κάναμε αυτό με το προσφυγάκι το 2005. και με την ε, ρέγγα του Ατλαντικού το 2007, του Βορείου Ατλαντικού. Είναι δυνατό και πρέπει να το κάνουμε τώρα και με το Σαφρίδι. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Άιζες, ξέρουμε ότι το σαφρίδι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και μπορούμε να ξεπεράσουμε τα επόμενα χρόνια ε, τα αλλιεύματα και να φτάσουμε σε ύψος 600.000 τόνους και παραπάνω. Η βιομάζα του, του σαφριδιού, επίσης από, τα στοιχεία που έχουμε, ε, πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν μπορούμε να καταλήξουμε ακόμα πουθενά και πρέπει να προωθήσουμε την έρευνα για αυτό το θέμα. Είναι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συμμετείχε στην φετινή έρευνα για το οικοσύστημα και ελπίζω ότι θα μπορέσετε και θα θελήσετε να συμμετάσχετε στο μέλλον σε αντίστοιχες προσπάθειες. Η καλή κατάσταση του αποθέματος του σαφριδιού είναι ενθαρρυντική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να χαλαρώσουμε τις προσπάθειες. Χρειαζόμαστε μία συμφωνία, μία ρύθμιση μεταξύ των παράκτιων κρατών για να μην φτάσουμε μία στιγμή που θα το μετανιώσουμε. Να μην φτάσουμε σε μία στιγμή που θα το μετανιώσουμε. Αλλιώς όλοι θα είμαστε υπεύθυνοι γιατί θέτουμε εν κινδύνο αυτό το απόθεμα που είναι τόσο πολύτιμο για την αλληλεία μας. Και βεβαίως είναι ακόμη πιο πολύτιμο για τη δική μας αλληλεία στα νησιά Φαρόε. Για να είμαι ρεαλιστής θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα χρειαστούν ένας ή δύο γύροι διαπραγματεύσεων απλώς. Θα χρειαστούν παραπάνω πρέπει να εξετάσουμε όλε τι εναλλακτικέ λύσει και να λάβουμε υπόψη μα τα διαφορετικά συμφέροντα των μεν και των δε. Είμαστε το ένα από τα τέσσερα παράκτια κράτη. Και ω τέτοιο σας διαβεβαιώνω ότι είμαστε δεσμευμένοι για να βρεθεί μια ισορροπημένη και διαφανής νέα ρύθμιση που θα εξασφαλίσει μια βιώσιμη ύπαρξη του σαφριδιού στο βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό. Το παιδάκι με το κόκκινο είναι ο γιος μου. Του αρέσει να ψαρεύει. Εμείς λέμε ότι το άχθος βαραίνει όλους μας. Όλους, πραγματικά. Ούτως ή άλλως, δεν κληρονομήσαμε το σαφρίδι από του προγόνου μα. Απλώ το δανειζόμαστε από τα παιδιά μα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ ειλικρινά που ήρθατε εδώ. Υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι σαφές και μου φαίνεται πολύ καλό το γεγονός ότι ήρθατε εσεί εδώ να μα εκφράσετε τις απόψει σα και να συζητήσετε και με τους ευρωβουλευτέ μας. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στους συναδέλφου Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριο Στίβενσον, τον οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Νίκλεσεν για την παρουσίασή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ διότι δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήρθατε εδώ σήμερα, διότι το γεγονός ότι η συνάδελφό σας από την Ισλανδία δεν δέχτηκε την πρόσκλησή μας, μάλλον ε, λέει κάποια πράγματα. Στη συνάντηση που είχαμε στα νησιά Φερόε στο παρελθόν, να πω δε εδώ ότι είχα πάει και στην Ισλανδία και είχα συναντήσει και υπουργού εκεί, αλλά όχι για το θέμα του Σαφριδίου. Και νομίζω ότι δημιουργείται γενικότερη εντύπωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι τα νησιά Φεροέ επιθυμούν, όπως μόλις μας είπατε κι εσείς, να βρουν μια ισότιμη συμφωνία για το θέμα αυτό. Δυστυχώς ε, δεν συμβαίνει το ίδιο όταν συζητάμε την κατάσταση του Αφριδίου με την Ισλανδία. Ελπίζω να κάνω λάθος και ελπίζω οι συζητήσεις που είναι εξελίξει στο Λονδίνο σήμερα να με διαψεύσουν διότι πραγματικά θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να είναι και η Ισλανδία ε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να ε, συμφωνήσει και αυτή και να δεχτεί τη συμφωνία για τα παράκτια κράτη. Όταν επισκέφθηκα πρώτη φορά τα νησιά Φερό, διαπίστωσα πόσο όμορφο είναι το μέρος αυτό και νομίζω ότι οι φωτογραφίες είναι και μια διαφήμιση και ενθαρρύνει τα μέλη της Επιτροπής να επισκεφθούν τα νησιά Φερό. Ε, κάτι το οποίο σας προτείνω και εγώ να κάνετε γιατί είναι εκπληκτική ομορφιά στο μέρος. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε ε, φέτος. Η βιομάζα του αποθέματος αναπαραγωγής ε, εκτιμάται το 2010 από τον ISIS ότι βρίσκεται στα 2,2 εκατομμύρια τόνους. Είχαν ε, θέσει όριο στους 570.000 ε, τόνους. Η αρχική συμφωνία με την Ισλανδία διότι πριν από 5-6 χρόνια η Ισλανδία εκφόρτωνε περίπου 350 ε, τόνους, χιλιάδες τόνους ε, ε, σαφρίδι. και είχαν ανέβει στους 2.000 ενώ φέτος είναι στους 130.000 τόνους, ε, ίσως και περισσότερους. Ενώ εσείς ε, στα νησιά Φερόεν είχατε 15.000 τόνους ετησίως, λιγότερο από το 5% του συνολικού ΤΑΚ και φέτος το αυξήσατε μόνο κατά 5.000 τόνους. Έχετε δίκιο λοιπόν όταν λέτε ότι συνεισφέρατε στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη και στην υγεία του Σαφριδίου, αλλά δυστυχώς έχετε συνεισφέρει λίγο διότι πρόκειται για μεταναστευτικό είδος και όπως ε, μας έδειξαν πολύ σαφώς και οι χάρτες σας, το απόθεμα του Σαφριδίου μεταναστεύει κάθε περίοδο από την ε, Ιβυρική Χερσόνησο, στην Ισλανδία και από εκεί στην ε, Ισλανδία, στα Νορβηγία και στα νησιά το Φαρόε. Και προσφάτω, λόγω της κλιματικής αλλαγής, πήγαν ακόμα πιο βόρεια και έφτασαν και μέχρι τα ύδατα της Ισλανδίας. Αλλά ο χρόνος στον οποίο παραμένει το σαφρίδι στα ύδατά σας είναι δύο μήνες το πολύ. Και ο χρόνος ο οποίος παραμένει σε ευρωπαϊκά και νορβηγικά ύδατα είναι περίπου εννέα μήνες. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές ενδείξεις ότι η υγεία και η ανάπτυξη του βιώσιμου αποθέματος συνδέεται περισσότερο με την ε, βιώσιμη αλία, κάτι το οποίο αναγνωρίζει και το MSC όπως γνωρίζετε. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταίροι μας στην Νορβηγία έχουμε αναλάβει ε, πολύ περισσότερα καθήκοντα, διότι εμεί είμαστε υπεύθυνοι και όχι εσεί για του δύο μήνε που παραμένουν τα αποθέματα στα δικά σας ύδατα. Υπάρχει το κατόφλι του ISIS των 570.000 τόνων για τη δική μας αλληλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Νορβηγία. Και επειδή το γνωρίζουμε αυτό, το να λένε τα νησιά Φερόες και η Ισλανδία ότι αφού θα υπερβούλα αυτή το δικό τους το ανώτατο όριο των 570.000 τόνων θα ε, αλλιεύσουμε και εμείς περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι ήταν μια αυθαίρετη απόφαση που επιδίνωσε το πρόβλημα. Και οδηγηθήκαμε σε μια κατάσταση όπου περίπου το 50% των εκτιμόμενων ε, ε, αποθεμάτων βιομάζα θα εκφορτώνονταν σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό θα ε, χαθεί το απόθεμα. Και ε, ναι μεν πολύ σωστά λέτε εσείς ότι εμείς δανειζόμαστε τα ψάρια αυτά από τα παιδιά μας. Επομένως κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι προς το συμφέρον όλων να βρούμε μια λύση, αλλά δεν μπορεί να είναι μια λύση η οποία απλώς θα ε, επιβραβεύει την αυθαίρετη συμπεριφορά των νησιών Φερόε και της Ισλανδίας φέτος. Ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή εσείς μπορείτε εύκολα να λιεύσετε 85.000 τόνους και η Ισλανδία 130.000 τόνους να μπορεί να υπάρξει ποσόστοση σε αυτό το όριο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει να γίνεται δίκαιη κατανομή των αποθεμάτων σε όλα τα παράκτεα κράτη και έτσι θα μπορέσει να είναι βιώσιμο και το είδος ε, για το μέλλον. Δεν θα πρέπει να καταστραφούν οι θέσεις ε, εργασίας των αλλιέων στο πελαγικό τομέα, στην Νορβηγία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι εξαρτώνται από αυτό το είδος εδώ και δεκαετίας και αυτή τη στιγμή τιμωρούνται ε, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών. Μπορεί να είναι προσωρινή η κατάσταση ε, για την παρουσία του αποθέματος ε, στα βορειότερα ύδατα της Ισλανδίας και των νησιών Φαρόε, αλλά μπορεί να αναστραφεί αυτή η κατάσταση και θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Ε, εάν αναστραφεί το τοπίο στα επόμενα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι θα βρεθεί ο πελαγικός μας τομέας σε πολύ μειονεκτική θέση. Είναι πολύ περίπλοκο το ζήτημα και σας ευγνωμονώ για άλλη μια φορά διότι κάνατε μια πολύ εύγλωτη και πολύ σαφή παρουσίαση και ουσιαστικά μας αποδείξατε για ποιον ακριβώς λόγο είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε συμφωνία μαζί σας ή δυνατόν και με την Ισλανδία. Αν δεν μπορέσουμε με την Ισλανδία δεν ξέρω τι θα γίνει αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ελπίζω επίσης η σημερινή μέρα να προσθέσει κάτι στην διάθεση που έχουμε όλοι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Από ό,τι φαίνεται και εσείς θέλετε να καταλήξετε σε συμφωνία μαζί μας και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο τώρα σε όλους όσους ζήτησαν το λόγο και από εκεί και πέρα θα σας δώσω και χρόνο για να απαντήσετε. Στη συνέχεια λοιπόν, η κυρία Ντότς. Thank you. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι που μετά από αρκετέ συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μπορούμε να μιλήσουμε στον οποίο και να σας εκφράσουμε τις απόψεις ε, των όσων εκπροσωπούμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε σήμερα και μας αφιερώσετε το χρόνο σας. Νομίζω ότι είναι ένα καλό βήμα προς τα εμπρός και το εκτιμούμε είναι ένα βήμα παραπάνω αυτό που κάνετε εσείς σε σχέση με όσα προτίθονται να κάνουν άλλοι. Όπως φαντάζεστε, αυτό το θέμα έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις μεταξύ των αλλιέων, των, οποίων οποίους εγώ προσωπώ, και από τη Βόρεια Ιρλανδία και από όσους... Is that um, και από τη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν που δουλεύουν στα σκοτσέζικα λιμάνια και σκέφτομαι μια συγκεκριμένη οικογένεια Ελίων από τη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουν επενδύσει τεράστια ποσά χρημάτων σε τελευταίες τεχνολογίες ε, εξοπλισμό σκεπτόμενοι ότι αυτή η συμφωνία που αναφέρεστε εσείς, στην οποία αναφέρεστε εσείς ως συμφωνία ad hoc, ξέρουμε ότι είναι μια ετήσια συμφωνία επαρακτήων κρατών και που θα συνεχιστεί και που θα βασίζεται στην, ε, σε συγκεκριμένες λογικές σκόπιμες διαπραγματεύσεις για το εγγύς μέλλον. Και δεν είναι μόνο για αυτούς σημαντικό, αλλά και για τους ε, πολίτες των νήσων Φερόε, και όσους ασχολούνται με το απόθεμα για τις γενιές των αλλιέων που θα έρθουν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και αυτό που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα για μας είναι ότι μονομερός κάποιοι έχουν αποφασίσει να δηλώσουν ε, την αύξηση στην ποσόστοση. Και αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό αντί να παραμείνουν δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να προσπαθήσουν να διεκπαιρεωθούν τα θέματα αυτά. Μιλήσατε για συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες, για όλα τα διαχειριστικά θέματα. Αυτό το θέμα έχει ε, μπει στα πλαίσια της Συμφωνίας των Παρακτήων Κρατών, την οποία αναφέρεται ως Συμφωνία Ad Hoc. Και αυτή η συμφωνία τύχε αιτήσεις και κατάφεραν να συγκλίνουν οι απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων ε, μερών ώστε να υπάρχει μια σωστή διαχείριση του αποθέματος το οποίο βρίσκεται και σε κίνδυνο. Και κάτι άλλο που ήδη αναφέρθηκε, είπατε ότι οι πολίτες των ε, νήσων ήθελαν να αυξήσουν την ε, την ποσόστοση λόγω του ότι το απόθεμα παραμένει σε περισσότερο χρόνο στα ύδατα των νησών Φερόε. Αν όμως κάτι τέτοιο γίνει, τότε μάλλον θα πρέπει να, να δώσετε λιγο, μικρότερο μερίδιο από την ποσόστοση. Ε, μήπως αυτό γίνεται για το προσφυγάκι. Μονομερός αυξάνουμε ε, την ποσόστοση γι' αυτό και τα προβλήματα που απορρέουν και όχι ότι το. και δεν, μήπως αυτό δεν οφείλεται στο γεγονό ότι το απόθεμα έχει ε, καταρρεύσει και δεν μπορεί να λιευθεί. Και τέλος να πω ότι αναφέρεστε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και 60% ε, με 70% της, οικονομικής, της οικονομίας των ΦΕΡΟΕ βασίζεται στην αλία. Κατανοούμε τους λόγους που συμβαίνει αυτό, την απομακρυσμένα το νησί, και πόσο σημαντικό είναι, πόσο σημαντική είναι η αλληλεία και για τις κοινότητες αλλά και για την οικονομία. Αλλά στενή συνεργασία και πρόσβαση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ευθύνη και από εσάς. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας σε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται. Χαίρομαι που ήρθατε. Ε, είναι πολύ ενθαρρυντικό που γίνονται συζητήσει έστω και σήμερα. Ε, αλλά πρέπει να πω ότι πρέπει να βρεθεί μια ισότιμη λύση για όλους. Δεν νομίζω ότι η μονομερής αύξηση της ε, ποσόστοσης είναι ισότιμη λύση. Ευχαριστώ. Ο Υπουργό θα μείνει μέχρι τις 12 μου είπαν. Επομένως θα ήθελα να σας ζητήσω να είστε λίγο πιο σύντομη για να μπορέσει να απαντήσει σε όλους σας. Η κυρία Άντρες Μπαρέα στη συνέχεια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό που ήρθε και μας εκφράζει τις απόψεις του εδώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, διότι εσείς μας είπατε ήδη ότι η αλλαγή του κλίματος σας έχει ουσιαστικά θέση στο επίκεντρο της αλίας του Σαφριδίου. Βρίσκεστε περικυκλωμένη από ψάρια και έχετε δυνατότητες αλίας. Οι επιστημονικές ενδείξεις όμως και ε, οι ποσοστώσεις που βγάζετε για κάθε χρόνο γίνονται από εσά ή ε, χρησιμοποιείτε και τα στοιχεία του ISIS. Από ποιον βγαίνουν οι ποσοστάσεις. Επίσης ακούσαμε ότι υπήρχε πρόβλημα επειδή δεν υπήρχε συμφωνία με τα παράκτια κράτη. Ποια είναι τα αίτια, τι ευθύνη έχει κάθε κράτος μέλος. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει καλή διαχείριση και δεν συμφωνούν τα παράκτια κράτη σημαίνει ότι ο καθένας καθορίζει τη δική του ποσόστοση και επομένω υπάρχουν ε, ε, μεγάλα προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι κάνει το κάθε κράτος. Ευχαριστώ κύριε Λεβίν. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Α, εδώ είμαι μπροστά σας, απέναντί σα αν με ψάχνετε. Κύριε Νίκλασεν, είναι πραγματικά κρίμα που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ο καθένας αποφασίζει τι ποσόστοση θα πιάσει ε, και ψαρεύει και ψάρια που ψάρευαν προηγουμένως άλλες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτεί. Και πρέπει να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο ψαρεύουν και διάφορες άλλες χώρες, όχι μόνο εσείς, αλλά αναπτυσσόμενες χώρες γιατί εμείς έχουμε συμφέροντα, αληφτικά συμφέροντα, ε, στα ύδατά τους. Μπορούμε τα ιστορικά αλλιεύματα να τα συζητήσουμε και να λάβουμε υπόψη. Εμείς οι πράσινοι θεωρούμε ότι αυτά τα αλλιευτικά δικαιώματα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και θα πρέπει να πάνε σε αλληλείς που ψαρεύουν βιώσιμα και περιβαλλοντικός πώς και λαμβάνοντας υπόψη της απασχόλησης. Μία ερώτηση κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι το 50% των αλλιευμάτων του σαφριδιού στα νησιά Φαροέ ε, προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και διατροφή. Είναι ένα θαυμάσιο ψάρι για την ανθρώπινη διατροφή. Θα ήταν λοιπόν σκάνδαλο να το, να προορίσουμε για πουθενά, για, για κάπου αλλού. Στην Ισλανδία, ας πούμε, Ξέρω ότι ψαρεύουν ε, το σαφρίδι για να θρέψουν τους ε, σολομούς της δατοκαλλιέργειας. Είναι σκάνδαλο για μένα. Το θέμα είναι λοιπόν, το σαφρίδι ας πούμε, τι θα το κάνουμε, θα το ψαρεύουμε για να το τρώμε εμείς οι άνθρωποι ή θα το κάνουμε ηχθιάλευρο μετά για την υδατοκαλλιέργεια. Αυτό είναι το, το ερώτημά μου. Εσείς πώς, πρέπει, πώς πιστεύω ότι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε το σαφρίδι. Η ε, κυρία Πατραγωνέβες. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Υπουργό που είναι σήμερα εδώ παρόν για να μιλήσει μαζί μας για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Μιλήσαμε και για την Ισλανδή Υπουργό. Στην δική σας παρέμβαση θέσατε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ότι δηλαδή θα πρέπει από κοινού να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και από κοινού να βρούμε μια λύση. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να συνέλθουν ώστε να μπορέσουμε όλοι να υποφεληθούμε. Μου άρεσε ιδιαίτερος αυτό που είπατε ότι δηλαδή είναι απαραίτητο όλοι μαζί να καταφέρουμε να σκεφτούμε ένα σχέδιο για την ευρωπαϊκή διαχείριση των αποθεμάτων. Τώρα ε, φτάσαμε σε κάποιες μονομερείς συζητήσεις. Ε, αποφάσεις βέβαια αυτές ε, προφανώς ε, θα πρέπει να εκλείψουν. Θα πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτούμε και να δούμε τι ακριβώς γίνεται και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί καταλήξαμε στην μετανάστευση των αποθεμάτων του Σαφριδιού. Και αυτό επίσης το είπε και ο συνάδελφος Στίβενσον. σε ποιο βαθμό η παρούσα κατάσταση είναι περιορισμένη χρονικά, θα συνεχιστεί, είναι κάτι παροδικό. Εδώ είναι απαραίτητο να υπάρξουν ε, και επιστημονικές ε, επιστημονικά στοιχεία ως προς αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει μια αξιολόγηση των φυσικών και χημικών παραμέτρων του νερού ε, και σε σχέση με μια περαιτέρω κλιματική ελλαγή. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς τώρα. Δεν υπάρχει όμως κάποιο συγκεκριμένο επιστημονικό πλαίσιο το οποίο να μπορεί να μας πει μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα εξελιχθεί περαιτέρω, τι γίνεται με, τα, με την αλληλεία των αποθεμάτων. Θα αυτό που συμβαίνει τώρα με το Σαβρίδι θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλα αποθέματα. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό αυτό είναι ένα δείγμα ή ένας δείκτης για αποφάσεις που θα πρέπει ίσως να ληφθούν για, σε, για παρόμοιες καταστάσεις που θα συμβούν σε άλλα αποθέματα. Υπάρχουν δηλαδή διάφορα είδη ανησυχιών που ας πούμε η ζωή των, των, των παρακτήων κοινοτήτων, ε, πώς θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται οι αλληλείς που έχουν παράδοση αλληλείας εδώ και εκατοντάδες χρόνια σε, τέτοια, σε τέτοιες κοινότητες. Όλα αυτά λοιπόν αυτή τη στιγμή διακυβεύονται. Και ε, οι άνθρωποι έχουν να αντιμετωπίσουν και την μετανάστευση των αποθεμάτων, που ίσως να είναι και κάτι προσωρινό. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Η κοινότητα των ε, αλλιέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να εξαρτάται από τη μετανάστευση, από τις μεταναστευτικές ροές των διαφόρων αποθεμάτων και των διαφόρων ειδών. Εδώ υπάρχει ανάγκη για επιστημονικές μελέτες. Δεν μιλούμε δηλαδή μόνο για την καταγραφή τάσεων, ε, μιλούμε για κάποιες μεσοπρόθεσμες προοπτικές. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι συγκεκριμένα οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες αυτών των ε, μεταναστεύσεων. Γιατί πλήττονται οι αλληλείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως ε, αύριο να πληγούν και οι αλληλείς οι δικοί σας. Και κάτι τελευταίο. Εγώ ήμουνα εισηγήτρια στην έκθεση του Κοινοβουλίου για τη μεταρρύθμιση της κοινή ελευτικής πολιτικής και εκεί στην έκθεση αυτή πάντα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση, θα πρέπει να, να υπάρξει περιφερειοποίηση των διαχειριστικών αρχών. γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό οι διάφορες περιφερειακές αρχές να έχουν ε, λόγο στη διαχείριση των αποθεμάτων τους. Υπάρχουν ε, διάφορα είδη τα οποία μεταναστεύουν προς τις ε, νήσους Φερόε ας πούμε. Είναι σαφές ότι η αλληλευτική προσπάθεια που καταγράφεται σήμερα με τα τάκια της προσωστώσης μπορεί να οδηγήσει στο ότι κάποια αποθέματα θα εξαφανιστούν και αυτό θα πλήξει ακόμη περισσότερο άλλα είδη α, ψαριών. Ε, εντάξει, αυτό ίσω να είναι λίγο δευτερεύον ερώτημα σε σχέση και με αυτό που είπε ο Υπουργό, αλλά ήθελα έτσι, αφού έχω το λόγο, να το αναφέρω ακροθυγώς για να, να μπορέσουμε να συζητήσουμε περαιτέρω για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις και σε όλα τα σχόλια τα οποία διατυπώθηκαν. Έχετε όσο χρόνο θέλετε στη διάθεσή σας. Εσείς ξέρετε ε, ότι πρέπει να φύγετε στις 12, επομένως έχετε όσο χρόνο θέλετε εσείς στη διάθεσή σας και σας αφήνουμε από εκεί και πέρα, ε, θα σας αποδεσμεύσουμε να πάτε στις υπόλοιπε υποχρεώσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. για τα ερωτήματά σας. Ήθελα να είμαι σήμερα εδώ για να ακούσω και τις απόψεις σας και να μου πείτε τι ακριβώς πιστεύετε και να μπορέσω να απαντήσω και σε ερωτήσεις. Ο κύριος Στίβενσον ήρθε στις ε, νήσους Φερόε και κάναμε κάποιες συζητήσεις. Κάναμε μία διάσκεψη μάλιστα και το θέμα ε, της διάσκεψης ήταν πώς μπορούμε να μοιραστούμε τα πελαγικά είδη, τα πελαγικά αποθέματα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήταν ο κύριος Στίβενσον παρόν και όταν ζήτησε βεβαίω να συναντηθεί μαζί μου, φυσικά είπα ναι, γιατί εμείς στις νήσους Φερόε πιστεύουμε στο διάλογο. Πιστεύουμε στις διαπραγματεύσει. Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε. Ο κύριος Στίβενσον είπε ότι υπάρχουν ε, πολύ ωραίες ε, φωτογραφίες της, ε, στην παρουσίαση. Ε, είμαι και υπουργό τουρισμού, τι να κάνουμε. Οπότε αν θέλετε να έρθετε, βεβαίως είναι πανέμορφα τα νησιά μας. Αλλά βεβαίως δεν μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε σαφρίδια, ε, αυτό εννοείται. Πολλά τα ερωτήματά σας, ε, δεν ξέρω αν θα προλάβω να τα απαντήσω όλα, θα προσπαθήσω πάντως. Τι αναμένουμε, τι μέλη γενέστε, ένα είναι αυτό το βασικό ερώτημα. Όπως σας είπα, πιστεύω στον ε, διάλογο και στις διαπραγματεύσεις. Και έτσι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε μια, σε μια συμφωνία για το προσφυγάκι για το 2005, από το 2005. Μας πήρε 8 με 10 χρόνια για να καταλήξουμε σε εκείνη τη συμφωνία και προφανώς αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για οποιονδήποτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα καταφέραμε και όλα τα παράκτια κράτη είναι μέρη της συμφωνίας αυτής πλέον. Κάναμε και συμφωνία για τη Ρέγκα. Αλλά αυτή η συμφωνία κρατάει από το 2004, αν θυμάμαι καλά. Βεβαίως από τότε έχουν υπάρξει διάφορες κλιματολογικές αλλαγές και τα αποθέματα της ράγκας έχουν μεταναστεύσει. Μας πήρε τρία χρόνια. Το 2007 καταλήξαμε σε μια νέα συμφωνία για τη ράγκα. Και αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι νέα συμφωνία για το Σαφρίδι. Ναι, όντως έχουν υπάρξει αλλαγές. Το πρόβλημα με τα ψάρια όταν μιλάμε για τον βόρειο ανατολικό Ατλαντικό είναι ότι τα ψάρια κολυμπούν. Και όταν τα ψάρια κολυμπούν πάνε από τα ευρωπαϊκά ύδατα στα ύδατα τα δικά μας. Και μετά μιλούμε για συνδιαχείριση. Δεν θέλω όμως τώρα να επικεντρωθούμε στα κλιματολογικά, παρόλο που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Υπάρχει λοιπόν τώρα ένα απόθεμα σαφριδιού στα δικά μας ύδατα, μπορεί να είναι για 5 χρόνια, για 10 χρόνια και μετά να φύγει. Φυσικά είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και θέλουμε να είμαστε και λογικοί, ρεαλιστές. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τα αποθέματα. Και είμαστε υπεύθυνοι και για τους πολίτες μας. Και για να το μοιραστούμε όπως θα πρέπει, δεν θα πρέπει να αναρωτιόμαστε, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. Ο κύριος Στίβενσον είπε ότι το Σαφρίδι παραμένει στα δικά μας είδατα μόνο για δύο μήνες. Ναι, αλλά πριν δέκα χρόνια αυτό. Αυτό έχει αλλάξει. Τώρα όλο το χρόνο βρίσκονται, βρίσκεται απόθεμα σαφριδιού στα ύδατά μας. Μιλούσαμε για 30.000 τόνους, περίπου 5% δηλαδή του ΤΑΚ. Και το δικό μας λογικό μερίδιο είναι 15% θεωρούμε. Γι' αυτό βάλαμε την ποσόστοση στους 85.000 τόνους. Αλλά πιστέψτε με, αν βάλουμε την ποσόστοση στους 200.000 τόνους δεν θα έχουμε πρόβλημα να το αλλιεύσουμε, αλλά δεν μιλώ γι' αυτό. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι τι υπάρχει σε, από πλευράς ε, επιστημονικών ε, αποτελεσμάτων. 15% είναι ένα λογικό και δίκαιο μερίδιο για μας. Φυσικά πρέπει να κάνουμε περισσότερη έρευνα. Φυσικά χρειαζόμαστε περισσότερα ε, επιστημονικά στοιχεία για το σαφρίδι. Και γι' αυτό εγώ ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να από κοινού και με την Ισλανδία και με την Νορβηγία και με, και εμάς να εμπλακεί στις διάφορες έρευνες για το βόρειο τμήμα του βόρειο-ανατολικού Ατλαντικού, διότι εκεί χρειαζόμαστε τα επιστημονικά στοιχεία. Επίσης, ένα ερώτημα τέθηκε που είπατε ότι μονομερώς θέσαμε τις ποσοστώσεις. Δεν έγινε έτσι. Αλλά εντάξει, εδώ μπορούμε τώρα να κάτσουμε και να κατηγορούμε ένα τον άλλον. Αυτό που έγινε ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Νορβηγία έθεσαν τις ποσοστώσεις τους. Αν πάρουμε την Νορβηγία και τις αυτές τις ποσοστώσεις, συνολικά ήταν παραπάνω από, την, από τις ποσοστώσεις που είχε θέσει η ISIS. Μόνο με αυτές τις δύο ε, μόνο με αυτή τη μία μάλλον διμερή συμφωνία το Σαφρίδι δεν ήταν πια βιώσιμο. Μόνο με τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας. Αλλά εμείς θεωρούσαμε, ε, σα είπα και πάλι ότι πιστεύουμε στις διαπραγματεύσει. Η Ισλανδία μετά από την διμερή αυτή συμφωνία έθεσε τη δική της ποσόστοση. Και κατά την άποψή μας ήταν αρκετά υψηλό η ποσόστοση που έθεσε. Μετά από αυτό έθεσε τη δική της ποσόστοση στα διεθνή ύδατα η Ρωσία. Και επίσης και η Ρωσία αύξησε την ποσόστοσή της. Τότε εμεί δεν είχαμε θέσει ακόμη ποσόστοση. Ο υπουργό Αλία μα προσπάθησε άλλη μια φορά να πάει στους διάφορους υπουργού Αλίας στα, των παρακτήων κρατών, Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Ισλανδία και να προσπαθήσει με κάποιο τρόπο να καταλήξουμε σε μια λύση. Αλλά δεν κατάφερε. Τώρα εμείς θέσαμε τη δική μας ποσόστοση και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, αλλά εν πάση πρέπει όλοι να σεβόμαστε όλους. Να δούμε ποιε είναι οι, επιστημονικές μελέτες και να μοιράσουμε τα πράγματα δίκαια. Ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες μας μπορούν να ζήσουν από αυτό τον πόρο που βρίσκεται στη... στα ύδατά τους. Οπότε εγώ εύχομαι να μπορέσουμε να κάνουμε πολύ περισσότερες επιστημονικές έρευνες από κοινού, να συνεχιστούν και οι διαπραγματεύσεις σήμερα που ήδη ξεκίνησαν στο Λονδίνο και εγώ από τη δική μας πλευρά μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Ακόμη και αν δεν καταλήξουμε σήμερα σε αποτέλεσμα στο Λονδίνο, Ελπίζω να γίνει αυτό στην επόμενη ή στη μεθεπόμενη συνάντηση. Μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Είμαι επιπισμένο. γιατί δανειζόμαστε το απόθεμα του σαφριδιού από τα παιδιά μας και το βάρος που έχουμε θα πρέπει να, μας, ε, να σταματήσει τις αλληλοκατηγορίες και θα πρέπει να δώσουμε τα χέρια ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο αποτέλεσμα, σε ένα δίκαιο μερίδιο για όλους. Ε, Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Γκάλαγκερ είχε ζητήσει το λόγο και χρειάστηκε να λείψει για λίγο. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, είχα πει ότι δεν θα δώσω το λόγο σε κανέναν άλλον, αλλά ε, αν εσείς μπορείτε να του μιλήσετε, θα, να το απαντήσετε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλαγκερ. Κύριε Γκάλαγκερ, θέστε την ερώτησή σας και τελειώνουμε με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χρειάστηκε να φύγω, ζητώ συγγνώμη. Ε, σε μία συνεδρίαση. Ε, την επόμενη εβδομάδα πάλι για, τον, για το Σαβρίδι θα μιλήσουμε. Έρχομαι τώρα από την Αλάσκα και επίσης ε, η εκλογική μου περιφέρεια ενδιαφέρεται πολύ για το Σαφρίδι. Ελπίζω να τελεσφορήσουν οι συζητήσεις στο Λονδίνο και να εξασφαλίσω μια, ένα βιώσιμο αλίευμα. Γιατί εσείς μιλήσατε για τις ε, μελλοντικέ γενιές και είναι σημαντικό να τους εξασφαλίσουμε τα αποθέματα. Αναγνωρίζω ότι τα νησιά Φερόε θα πρέπει να πάρουν κάτι παραπάνω και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να τα υποστηρίξει. Τώρα, αν θα τριπλασιαστεί ή τέτραπλασιαστεί η ποσόστοση, αυτό είναι θέμα συζήτησης. Αλλά το απόθεμα είναι ενιαίο και δυστυχώ το πρόβλημα είναι ότι όλα τα παράκτια κράτη δεν το αναγνωρίζουν αυτό. Οι επιστήμονες μας λένε ότι μόνο το 0,7% του αποθέματο είναι στα νησιά Φερόε. Δεν ξέρω αν το δέχεστε αυτό. Γιατί κινείται το απόθεμα και αλλάζει. Όταν έγινε αυτή η επισκόπηση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, οι επιστήμονες μας είπαν πέρυσι ότι το ΤΑΚ θα έπρεπε να είναι στα 560, 560.000 τόνους. Ενώ στην πραγματικότητα το ΤΑΚ έφτασε πάνω από τις 700.000 τόνους. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Από ό,τι ξέρω εγώ από την ε, Αλία, η τιμή του ψαριού εξαρτάται από την ποσότητά του. Από την ποσότητα που εκφορτώνεται. Αν όλοι σεβαστούμε το τάκ και τις ποσοστώσεις μας, τότε νομίζω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια καλή τιμή για τους ε, ε, ψαράδες μας. Αν πουλιέται όμως ε, στη μαύρη το ψάρι, τότε οι τιμές πέφτουν. Και ελπίζω όλες οι χώρες να σεβαστούν αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ελπίζω οι δικοί σας αξιωματούχοι και οι δικοί μας και οι Ισλανδοί αξιωματούχοι. Έχω πάει πρόσφατα στην Ισλανδία και γνωρίζω πολύ καλά ε, τις απόψεις του Υπουργείου Αλίας της Ισλανδίας. Και ελπίζω να μην αυξήσουν ε, τα τάκ και στην Ισλανδία. Ε, ελπίζω λοιπόν όλοι να σεβαστούν ε, τα νούμερα. Δεν πρέπει να μιλάω σαν επιστήμονας, θα πρέπει να προσέξω πώ θα μιλήσω. Έχουμε ένα μνημόνιο ενημερωτικό. Έχω φέρει πολλά αντίτυπα. μπορείτε να πάρετε κάποιο, αν σας ενδιαφέρει, για να δείτε τη θέση των νησιών Φερόε. Λέτε το 0,7% είναι στα δικά μας ύδατα. Αυτό είναι το συνολικό νούμερο. Το 2007 είχαμε αυτή την επισκόπηση και φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που συμμετείχαμε στην επισκόπηση αυτή του Ινστιτούτου. Και αν δεν απατώμε, για πρώτη φορά ε, λάβουμε υπόψη μας όλη την περιοχή των Φερόε. Μέχρι τώρα όλοι πίστευαν ότι το Σαφρίδι είναι πιο νότια και έτσι ήταν, αλλά το πράγμα άλλαξε. Το Θαλάσσιο Ερευνητικό Ινστιτούτο των Φερόε έχει κάνει και άλλες ε, μελέτες οικοσυστημάτων ε, και προς την Νορβηγία και προς την Ισλανδία και μας ε, δίνει μια τελείως διαφορετική εικόνα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά και οι επιστήμονες ακόμη αναγνωρίζουν ότι έγινε μεγάλη αλλαγή του πώς κινείται τελείως διαφορετικά και βρίσκεται σε τελείως άλλο χώρο πλέον το απόθεμα στα φρυδιού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα επιστημονικά στοιχεία. Τώρα, εμείς από πλευράς μας οι πολιτικοί δεν πρέπει να καθόμαστε και να συζητάμε αν το απόθεμα είναι 0,7% ή 15% όπως ανέφερα. Το θέμα είναι να συζητήσουν οι επιστήμονές μας. Να κάνουν ε, μελέτες οικοσυστημάτων, μελέτες ε, γόνων στο Βόρειο Ατλαντικό και να συμπεριλάβουν όλα τα σημεία όπου βρίσκεται σαφρίδι. Ούτως ώστε να δούμε ποια είναι η πραγματική εικόνα και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Πέρυσι η ποσόστοσή μας ήταν 30.000 τόνους και φέτος 85.000 τόνους. Υπήρξε αύξηση, όντως. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε με την Νορβηγία και η Νορβηγία μπόρεσε να ψαρέψει 70.000 τόνους περισσότερους από την πέρυσι. Και λέει ότι το κάνουν αυτό επειδή πέρυσι δεν ψάρεψαν. Αυτό είπε η Νορβηγία. Επομένω, δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση την αύξηση τη ποσότητα τη Νορβηγία κατά 70.000 τόνου. Αυτά που άκουσα εδώ και από τι διαπραγματεύσει, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να δεχτεί μια αύξηση τη της ποσότητας των Φερόε από τις 30.000 στις 85.000. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο διάλογος είναι καλύτερη λύση, η διαπραγματεύση είναι καλύτερη λύση. Και πιστεύω ότι ως πού θα φτάσουμε σε συμφωνία. Μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλα τα μέρη, γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Αν πετύχω μια συμφωνία όπου κάποιες χώρες ε, θα είναι μη ικανοποιημένε, θα τις ρίξουμε δεν νομίζω ότι θα είναι σόφρον. Πριν από δύο εβδομάδε ε, στο Λονδίνο ήταν καλέ διαπραγματεύσει. Ε, υπήρξαν μετακινήσει θέσεων, ε, κατανοήσαμε η μεν τη θέση των δε. Και χαίρομαι που συνομιλούν πολύ ήρεμα και συνομίλησαν πολύ ήρεμα στι τελευταίε διαπραγματεύσει η δική σα και οι δική μα. Ελπίζουμε ότι οι σημερινέ και αυριανέ διαπραγματεύσει θα μα οδηγήσουν κάπου. Γιατί χρειάζεται μια λογική συμφωνία. Χρειάζεται μια νέα μορφή διαχείρισης και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την επιτύχουμε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ εξ ονόματος όλων των συναδέλφων για την παρουσία σας και για την ε, διάθεσή σας να συζητήσετε με όλους εμάς. και ελπίζω όλοι να καταλήξετε σε συμφωνία και να μην φτάσουν ε, να περάσουν 10 χρόνια για να καταλήξουμε σε μια διμερή συμφωνία. Ε, θέλουμε μια συμφωνία που θα λαμβάνει υπόψη ε, την ε, αλληλεία, βιώσιμη για όλους και ελπίζω και τα δικό σας τα παιδιά αλλά και τα δικά μας να συνεχίσουν να αλληλεύουν. Ευχαριστώ πολύ. you,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 Να συνεχίσουμε τώρα γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει την ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η καταπολέμηση τη παρόμοιη σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έκθεση πρωτοβουλίας που ζήτησε η ομάδα των Πρασίνων, η συγγήτρια κυρία Λεβίν και να της δώσω λοιπόν το λόγο χωρίς περιττέρω καθυστέρηση για να μας πει κάποια πράγματα για την έκθεσή της. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που η Επιτροπή αποφάσισε να ε, κάνουμε αυτή την έκθεση για να δούμε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην καταπολέμηση παράνομης ελίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως γνωρίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περάσει πολύ σημαντικούς κανονισμούς, ε, κανονισμούς ελέγχου και επίσης υπάρχει και ο κανονισμός για την παράνομη λαθρέα και άναρχη αλληλεία και φυσικά τα προγράμματα αδειοδότησης για την αλληλεία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί σημαίνει ότι έχουμε λάβει πολύ σημαντικά βήματα για να ε, προστατεύσουμε από την παράνομη αλληλεία. Αλλά ακόμα δεν έχει επιληθεί το ζήτημα φυσικά. Μπορεί να υπάρχει καλύτερη νομοθεσία εσωτερικά, αλλά θα πρέπει να δούμε και λίγο πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα για να δούμε πώς μπορούμε να επηρεάσουμε και σε διεθνές επίπεδο και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην καταπολέμηση της παράνομης Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, Έχουμε απώλειες ε, της τάξης των 23, 23 ε, δις ε, δολαρίων ετησιών και μιλάμε για 20 με 26 εκατομμύρια τόνους που αλλιεύονται παρανόμως ετησίως. Και αυτό είναι περίπου το 1 πέμπτο του συνολικού παγκόσμιου αλεύματος. Επομένως είναι τεράστιο το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός ε, παράγων όταν ε, συζητάμε την αλληλεία και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να διαδραματίσουμε και πιο ουσιαστικό ρόλο. Θα πρέπει να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Στην έκθεση θέλουμε να εξετάσουμε διάφορες ε, πτυχές στις οποίες θα μπορούσε να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ε, αντιμετωπίσουμε παγκοσμίως την κατάσταση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας. Επίσης, θέλουμε να κάνουμε μία απόπειρα ώστε να προωθήσουμε τον ε, κανονισμό ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των περιφερειακών οργανώσεων αλληλείας. Ε, επίσης, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και διαμέσου των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με κράτη που ε, πλοηγούν σκάφη με σημαίες ευκαιρίες και λιμένες ευκαιρίες. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διότι σε κάποιο βαθμό ε, οι περιοχές αυτές αποτελούν φορολογικούς παραδείσους και θα πρέπει να βρίσκονται στην ε, κορυφή των προτεραιοτήτων μας ώστε να αντιμετωπιστούν. Επίσης υπάρχει και το μακροχρόνιο πρόβλημα του πώς μπορούμε να έχουμε ε, μια κατάλληλη σχέση μεταξύ της σημαία και του σκάφους. Διότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο το οποιοδήποτε λιευτικό σκάφος να αλλάξει σημαία αν υπάρχει απειλή ε, για σύλληψη και κατάσχεση του σκάφους. Είναι πολύ εύκολο για τους πλειοκτήτες να αποκρύψουν την ταυτότητά του, ε, να έχουν κάποιον αντιπρόσωπο και να μην γνωρίζουμε ποιο είναι ο ίδιος ο πλειοκτήτη. Και αυτή η κατάσταση πρέπει να πάψει να υφίσταται. Ε, μίλησα με κάποιον Σουηδό Αλία, ο οποίος μου εξήγησε πόσο εύκολο είναι να αλλάξει σημαία ενό σκάφου και από Σουηδική σημαία να γίνει για παράδειγμα ε, μία σημαία ε, νησιών ε, άλλων πήγε στο διαδίκτυο και μέσα σε 20 λεπτά είχε αλλάξει σημαία. Και αυτή η διαδικασία της ε, πολύ εύκολης ε, αλλαγής σημαίας διευκολύνει την παράνομη θα πρέπει επίσης να δούμε και τι γίνεται με όλες τις αλληλευτικές συμφωνίες ε, και τις συμφωνίες εταιρικέ ε, σχέσεις και τμήμα των κονδυλίων που δίνονται σε αυτές τις συμφωνίες είναι ε, για να βοηθηθεί ο τοπικός πληθυσμός, ο τοπικός αλληλευτικός πληθυσμός. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει καλύτερο συντονισμός μεταξύ χωρών σε πιο απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου, να εξετάσουμε τα γενικότερα συστήματα και να βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, σημείων αυτών. Θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και θα πρέπει να δούμε και κάποιες τεχνικές λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν επίσης. Παραδείγματος χάρη μητρώα DNA, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξεταστεί στην Ίσπρα στο Κοινό Κέντρο Έρευνας ε, ε, στον τομέα της αλίας και επίσης θα δούμε, να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ε, παρακολούθηση μέσω δορυφόρου των σκαφών. όσον αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης, Υπάρχουν δύο έγγραφα εργασίας τα οποία θα παρουσιαστούν. Το πρώτο θα παρουσιαστεί στις 25 συγγνώμη, μεταξύ 25 και 27 Ιανουαρίου που θα παρουσιάζει μια συνολική εικόνα των διαφόρων μέτρων και κανόνων τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή στις διάφορες περιφερειακές οργανώσεις ε, αλίας. Ε, θα ασχοληθούμε με θέματα παράνομης αλίας, τι κυρώσεις είναι διαθέσιμες και τι καθήκοντα αναλογούν στα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της παράνομης αλίας και φυσικά τι δυνατότητες συντονισμού υπάρχουν ε, για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Επίσης, 15-16 ε, Μαρτίου θα παρουσιάσουμε και ένα δεύτερο έγγραφο το οποίο θα παρουσιάζει τις διάφορες μορφές τεχνολογίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας και επίσης υπάρχει και η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ελπίζουμε ότι θα είναι έτοιμη η έκθεση προς ψήφιση τον Ιούλιο του 2011. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πατράωνα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη προσοχή Άκουσα την ε, παρουσίαση της κυρίας Λόεβιν. Τα όσα ακούστηκαν πραγματικά πρέπει να τύχουν της προσοχής μας και βεβαίως ε, ανήκουν στο συνολικό θέμα που μας απασχολεί, την ε, παγκόσμια αντιμετώπιση της παράνομης αλίας. Ζήτησα το λόγο γιατί δεν κατάλαβα κάτι. Νομίζω Μιλήσατε για τα μητρώα των αποθεμάτων και το πέρασατε λίγο γρήγορα. είναι λίγο προβληματικό για μένα όλο αυτό το θέμα. Δεν θέλω τώρα βέβαια να αναφέρω όλες τις, όλα τα κανθόδη προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από αυτά τα μητρώα. Γιατί εξαρτάται και αυτό το, από το πώς θα παρουσιαστεί αυτό το μητρό. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει θέμα ιδιωτικής ζωής. Ε, οπότε εκεί ξεκινάμε με προσωπικά δεδομένα κλπ. Οδηγούμεθα σε τεράστια προβλήματα. Οπότε καλό θα ήταν να μας πείτε λίγα πράγματα περισσότερα. Θα πρέπει να ξέρουμε γενικώ τι γίνεται με τις πτυχές αυτού του θέματος. Τώρα, κάτι ουσιαστικότερο. Εάν κατάλαβα καλά, Τα περισσότερα θέματα που αναφέρετε έχουν να κάνουν με το ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνολογίες κινητές ώστε να αντιμετωπιστεί η ε, παράνομη αλληλεία. Ε, φυσικά είναι σημαντικό αυτό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα που ίσως να είναι εξίσου σημαντικό. Δηλαδή, οι ίδιοι οι αλληλείς θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί αυτοί θα είναι οι βασικοί παίχτες στο παιχνίδι αυτό για να αντιμετωπιστεί η α, παράνομη αλληλεία. Αν προσπαθούμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημα και να ελέγξουμε απ' έξω προς τα μέσα την παράνομη αλληλεία, μέσω ας πούμε χρήσης διαφόρων τεχνικών μέσων ε, ε, θα πρέπει πάντα να υπολογίζουμε ότι οι ε, αλληλείς είναι πάρα πολύ δημιουργικοί όταν θέλουν για να σπάσουν το σύστημα. Για να, αν θέλουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε την παρανομιαλία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μοντέλα και μεθόδους τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι ίδιοι αλληλείς γιατί και αυτοί είναι παίχτες στο, στο παιχνίδι αυτό. Έτσι, απλά κάποιες σκέψεις να έφερα, ίσως να αξίζει τον κόπο να τις δούμε λίγο περισσότερο και πολύ σύντομα να πω ότι υπάρχει δυνατότητα να δοθούν ε, επιδοτήσεις ανεξάρτητα από το αν οι αλληλείς είναι διατεθειμένοι να καταγράψουν τα αλλιεύματά τους για να έχουν ας πούμε την, ε, ε, για, να, για την, ε, αν δηλαδή τα σκάφη τους δεν, είναι, δεν αλλιεύουν παράνομα, τότε μπορούν να καταγράψουν τα αλλιεύματά τους. Ε, υπάρχουν κάποιες ρήτρε για τους βασικούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να συμπεριληφθούν και να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε επιτυχείς. Κλείνοντας, να μην ξεχνάμε ότι για την παράνομη αλληλεία θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις επιστημονικές αξιολογήσεις. Δηλαδή, ε, οι επιστημονικές αποδείξεις πολλές φορές δείχνουν ότι έχουν γίνει λαθασμένες καταγραφές των αποθεμάτων. Ευχαριστώ λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσει να μιλήσει και η Κομισιόν. Σύντομα, ότι χρειαζόμαστε ελέγχους για την παράνομη αλία, φυσικά συμφωνούμε όλοι. Είναι γι' αυτό ένα μέσο για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη αλία. Αλλά πρέπει να προσέχουμε ώστε να υπάρξουν και σαφή πλεονεκτήματα για τους αλληλείς που τηρούν τους κανόνες. Εάν ε, θεωρήσουμε όλους τους αλληλείς υποπτούς, αυτό είναι διεκριτική μεταχείριση. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί, δεν συνάδει και με τις αρχές μας. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα πολιτικό κίνητρο για αυτούς που τηρούν τους κανόνες να έχουν ένα επιπλέον ε, πλεονέκτημα έναντι όσων ε, δεν ε, τηρούν τους κανόνες. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ω μέλος της επιτροπή ανάπτυξη δεν θα σε εκπλήξει ότι θα θέσω το εξή ερώτημα. Θα ήθελα να μου πει η συγγήτρια τι συνεισφορά μπορούμε να έχουμε ε, στον αγώνα καταπολέμησης της λαθρέας άναρχης και παράνομης αλίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θα θέλει να πάρει το λόγο ή εσείς θέλετε πρώτα, η συγκήτρια. Εσείς, η συγκήτρια. Ευχαριστώ. Ξέχασα να σας πω ότι χάρηκα που συνεργάστηκε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ίσως ε, σε ό,τι αφορά τα μητρώα DNA υπήρξαν κάποιες παρεξηγήσεις. Στο κοινό ερευνητικό κέντρο στην Ίσπρα στην Ιταλία ε, μιλάμε για κάποια αποθέματα ε, ψαριών, ε, για τα νερά στα οποία ζουν, για να βελτιώσουμε την ιχνηλασιμότητα των αλλιευμάτων. Δεν μιλάμε για, για DNA και για μητρώα, DNA ε, ούτε των επαγγελματιών αλλιέων, ούτε των σκαφών. Σε καμία περίπτωση δεν υπενήχθηκα κάτι τέτοιο, έτσι. Ήθελα να σας το ξεκαθαρίσω αυτό. Επίσης, δεν θα εξετάσουμε μόνο τεχνικές λύσεις του προβλήματος. Η έκθεση προσπαθεί να δει τι, υπάρχουν, τι, τι, δομές υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και ποιες δομές μπορούν να βελτιωθούν ούτως ώστε να ενδυναμωθεί η συνεργασία μας και ούτως ώστε να έχουμε πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία και εκτός της Ευρωπαϊκής, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία Ρόιμε, η έκθεση αυτή δεν θέλει να κατηγορήσει κανέναν ψαρά, ούτε αυτούς που αδιαφορούν για τους κανόνες. Έχουμε ένα κανονισμό τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τέθηκε σε ισχύ και αυτό σημαίνει ότι αν χρειαστεί μπορούμε να έχουμε πολύ πιο αυστηρού ελέγχους των Ευρωπαίων αλλιέων, πολύ πιο αυστηρού από αυτού που υπάρχουν σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ε, διεθνώς ε, μεγαλύτερη ισοτιμία. Το 70% του ψαριού που καταναλώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα εισάγεται, προέρχεται από άλλε περιοχέ και χώρε. Επομένω, πιστεύουμε ότι εμεί στην Ευρώπη έχουμε συμφέρον, πολύ περισσότερο εμεί από άλλου, να εξασφαλίσουμε ότι τα ψάρια αλλιεύονται νόμιμα. Γιατί η παράνομη αλλία δημιουργεί ένα μηχανισμό dumping. Ε, γινόμαστε εμείς ε, χώρος dumping ψαριών. Ε, κάνει κακό στο περιβάλλον και δημιουργεί και αστάθεια παντού. Κοιτάξτε τη Σομαλία, τι γίνεται. Το πρόβλημα της, Σομα... της πειρατείας στη Σομαλία προέκυψε από τις δυσκολίες λόγω της απόλυτης ελεύθερης πρόσβασης στα ύδατα της Σομαλίας. Όλα τα έθνη και η Ευρώπη έμπαιναν εκεί πέρα και ψάρευαν επί πολλά χρόνια στα νερά της Σομαλίας χωρίς κανέναν έλεγχο. Και αυτό δημιούργησε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα με τους πειρατές. Οι πειρατές ξεκίνησαν κυνηγώντα τους παράνομους αλείς και προσπαθούν να τους διώξουν από τα νερά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει διεθνώς το πρόβλημα της παράνομης αλίας. Τώρα που ασχολούμαι πιο λεπτομερώς με το θέμα αυτό, βλέπω πόσο ενδιαφέρον είναι να καταλάβουμε ποια άλλα θέματα συνδέονται με την άναρχη παράνομη και ρύθμιστη αλεία ε, Ποια μέσα, ποια μέτρα υπάρχουν, τι, τι έχουμε στη διάθεσή μας για να την καταπολεμήσουμε. Αυτό που έχουμε δεν είναι πολύ αποτελεσματικό. Δεν ξαναγκάζουμε χώρες να, την, να εξερευνήσουν, να, την, να διώξουν, αν θέλετε, την, αυτή την αλεία Απλώς προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τους υπάρχοντες οργανισμούς και φορείς. Α, μία ερώτηση που έγινε από μία άλλη βουλευτή ήταν για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε για το πρόβλημα σε αυτές τις χώρες. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός για την εποπτεία και την παρακολούθηση. Αυτές οι χώρες δεν μπορούν να ασκήσουν παρακολούθηση και έλεγχο αποτελεσματικά. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη περιφερειακή συνεργασία. Και εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα σημαντικότερο ρόλο, να βοηθήσει τι αναπτυσσόμενε χώρε να βελτιώσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία του. Ευχαριστώ. Η Κομισιόνα μπορεί μέσα σε πέντε λεπτά να μα ε, σκιαγραφίσει μια σφαιρική εικόνα ε, της κατάστασης. Ε, Δυστυχώ δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα το ξαναζητήσουμε σε άλλη περίπτωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας. Μέχρι τούδε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα υπέρ της καταπολέμησης αυτής της αλληλεία. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημιουργήσαμε το νέο ε, μηχανισμό για τους ελέγχους και τον κανονισμό για την καταπολέμηση της παράνομης και άνορχη αλίας. Χαιρόμαστε για αυτή την πρωτοβουλία σας λοιπόν. Νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να βρούμε και νέες λύσεις. Όπως είπε η συγγήτρια, ε, το γεγονό ότι υιοθετήσαμε τον κανονισμό αυτό για του ελέγχου και την παράνομη αλληλεία δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε τη δουλειά μα. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε τον κανονισμό για του ελέγχου, τον κανονισμό για την παράνομη αλληλεία και όπω είπε και η συγγήτρια, να δραστηριοποιηθούμε σε διεθνέ επίπεδο, ούτω ώστε να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να εξάγουμε κάποιε καλέ ιδέε ε, που σκέφτηκε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καταπολέμηση της αλίας. Μιλήσατε για κίνητρα για τους επαγγελματίες ψαράδες. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σήμερα έχουμε τέτοια μέτρα, παύλα κίνητρα, στον κανονισμό για τους ελέγχους και για την παρανομή και χρήσιμο θα ήταν να εξάγουμε εντό αγωγικών ε, διεθνώ αυτέ τι ιδέε, ούτω ώστε οι ψαράδε που ψαρεύουν στα ανοιχτή θάλασσα ή αυτοί που συμμετέχουν σε περιφερειακού οργανισμού να συμμετάσχουν στην, ε, στην προσπάθεια αυτή, στον αγώνα αυτό. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που είπε η κυρία Στάινε είναι ότι δεν θέλουμε τώρα εδώ να κατηγορήσουμε τους ε, ψαράδες. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Όπως είπε η συγγήτρια, θέλουμε να υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των διαφόρων αλλιέων, όποια και είναι η εθνικότητά τους, όπου και αν ψαρεύουν, σε οποιαδήποτε νερά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σκεφτούμε πολλά ακόμα. Ε, Μπορούμε πολλά να κάνουμε σε επίπεδο συμβαλωμένων μερών και σε επίπεδο κρατών μελών. Θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσει όταν ε, εντοπίζουμε παράνομε δραστηριότητε. Άκουσα τον προηγούμενο μιλητή. Αναφέραμε περιπτώσεις υπεραλίευση. Φυσικά θα πρέπει να ε, επιβάλλουμε κυρώσει σε περίπτωση υπεραλίευση και στι περιφερειακές οργανώσεις αλίας θα πρέπει να προβλέψουμε μηχανισμό κυρώσεων αυτών των δραστηριοτήτων, των παράνομων, σε όλα τα επίπεδα. Ε, σε επίπεδο κράτους σημαίας, σε κράτους εισαγωγής και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν θα υπήρχε αγορά παράνομης αλίας αν δεν υπήρχε εμπορευματοποίηση παράνομων αλλιευμάτων. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πράγμα να το επενθυμίσουμε στους ε, περιφερειακούς οργανισμούς αλίας. Επίσης, δεν θα υπήρχαν ε, σημαίες ευκαιρία εάν δεν υπήρχαν οι ευκολίες που γνωρίζουμε. Η δυνατότητα που έχουμε για να αλλάξουμε σημαία σε σκάφος. Όπως είπατε, στο ίντερνετ για να αλλάξουμε σημαία αρκεί να πληρώσουμε 500 δολάρια, χωρίς κανέναν έλεγχο. Τσακ, αλλάζουμε σημαία. Νομίζω ότι με τη βοήθειά σας λοιπόν μπορούμε να παίξουμε πιο ενεργό ρόλο στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που ανέφεραν οι Ευρωβουλευτές σήμερα. Νομίζω ότι είναι μια θαυμάσια πρωτοβουλία. Η Κομισιόν θέλει να συνεργαστεί όσο μπορεί περισσότερο μαζί σας, γιατί είναι για το συμφέρον μας, όπως είπατε. Είμαστε οι πρώτοι παγκόσμια αγορά. Είμαστε η δεύτερη αλή παγκόσμια και επομένω έχουμε μια τεράστια ευθύνη σε αυτό το τομέα. Εγώ σας ευχαριστώ και με αυτό ολοκληρώθηκε το σημείο υπαριθμό 16. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε επόμενες συνεδριάσεις. Να περάσουμε λοιπόν στα διάφορα, σημείο 17 και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο συνάδελφο Πούνσκης μετά από πολλά χρόνια δουλειάς μαζί μας ε, μας ε, αφήνει λόγω κινητικότητας εδώ στο Κοινοβούλιο έκανε πολύ σημαντική δουλειά στη γραμματεία της Επιτροπής Αλίας και τώρα μεταφέρεται στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο ε, λυπούμαστε που φεύγει αλλά του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη νέα του Επιτροπή και τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε εδώ στην Επιτροπή Αλίας ευχαριστώ και καλή τύχη Αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο στα διάφορα, ο κύριος Φερέιρα, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε. Η συζήτησή μας για τις δημοσιονομικές προοπτικές ε, διεκόπη. Σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Ναι, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε μία άλλη μέρα. Ο κύριο Γκαρίγα μου άφησε ένα σημείωμα για τα όσα τον είχα ρωτήσει. Ζητώ συγγνώμη που δεν σα το διαβίβασα. Θα συνεχίσουμε όμω τη συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση. Ε, δεν θα έχουμε και χρόνο άλλωστε τώρα να το συζητήσουμε. Ο κύριο Γκαρίγια ήρθε, έπρεπε να φύγει, έπρεπε να δώσουμε προτεραιότητα στον Υπουργό, δεν γινόταν αλλιώ. Θα προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε το σημείο στην ημερήσια διάτυξη σε μία από τι επόμενε συνεδριάσει και σα ευχαριστώ που μου το υπενθυμίσατε. Συγγνώμη που δεν το εξήγησα. Τώρα, έχουμε στο 18 τις ανακοινώσεις Προέδρου για τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Εγκρίνονται οι αποφάσεις, αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση. Και τώρα, ημερομηνία και διεξαγωγή της προσεγού συνεδρίασης 8 Νοεμβρίου 3 ε, με 6.30 και 9 Νοεμβρίου 9 με 12.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς Πρόεδρος. Πέρασε συνεδρία.